να διοριστεί μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Επιστημικής Ασφάλειας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Δεν βλέπω αντιρρήσεις, οπότε αυτός ο διορισμός ε, επικυρώνεται. Να περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου.